Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά στην προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα χαλιβουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Αμαλία Σαρτόρη, συντάκτης της προφορικής ερώτησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φρονώ ότι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έγινε μια συζήτηση για τα θέματα της βιομηχανίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης που όπως μας υπενθύμησε ο Επίτροπος μόλις προλίγο ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Κάναμε συζήτηση στην αίθουσα με τον Επίτροπο Άντορ και τον Επίτροπο Ταγιάννη και συνεχίστηκε γιατί μετά μιλήσαμε για την ενέργεια επιμακρών Αναφερθήκαμε επίσης στα προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας και συνεχίζουμε τώρα με την ερώτηση την οποία έθεσα εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας και θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα εδώ. Μας καθησύχασαν μάλιστα και ότι θα υπάρχει ένα ψήφισμα το Δεκέμβριο επί του ζητήματος και θεωρώ ότι όλα όσα ε, ψηφίσαμε χθες στην αρχή της ε, συνεδρίασης ε, βοηθά να ενισχύσει ε, την φροντίδα που δείχνει το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. υπάρχουν αρκετές βιομηχανικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το χάλιβα, ε, το σίδερο, τα σιδηρομεταλλεύματα και φυσικά βοηθάει και όλες τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Πρωτίστως στην αυτοκινητοβιομηχανία, ε, τη μηχανική, τον κατασκευαστικό τομέα, τους αγωγούς, ε, μεταλλικά εμπορεύματα, καθώς επίσης και στην αυτο, ε, ε, στα είδη χρήση ηλεκτρικά είδη, καθώς και άλλα. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν τομέας για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Το 2000 ε, η Ευρώπη έχασε την πρωτιά της και παραχώρησε την ε, πρώτη θέση στην Κίνα και τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη επέλεξε να επενδύσει πολύ σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρόκειται βέβαια για μια επιλογή την οποία συμμεριζόμαστε κι εμείς, αλλά αυτό είχε κατα... Ε, ως συνέπεια να μειωθεί η παραγωγή στον τομέα αυτό, αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκε και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ε, στην Ευρώπη η ηλεκτρική ενέργεια στοιχίζει 100% περισσότερο από ό,τι ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και για κάποια ε, κράτη-μέλη είναι σημαντικό και το κόστος του χρήματος. Τα τελευταία ε, χρόνια και το, τους τελευταίους μήνες φτάσαμε στα μέγιστα ιστορικά. Το 2007-2008 είχαμε μία μείωση κατά 16% στις θέσεις εργασίας στη Χαλιβουργία και σήμερα είμαστε στις 163 ε, κατασκευαστικές μονάδες. Υπάρχουν επίσης τεράστιες απώλειες και για το 2012 και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι υπάρχει πολύ σημαντική μείωση στην παραγωγή σε τομεί που σχετίζονται στενά με την ε, χαλιβουργία, δηλαδή αυτοκινητοβιομηχανία και κατασκευαστικό τομέας, που μόνο το 2011 είχαν μείωση της παραγωγής τους κατά 3,2%. Οι εξαγωγές αυξάνονται και φυσικά το διοικητικό άθος το οποίο βαραίνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει και επιπλέον κόστος που σημαίνει ότι μειώνονται οι δυνατότητες επενδύσεως στην καινοτομία και στην έρευνα και ευνοούν τις ξένες χαλιβουργίες. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε μήπως με τη νέα πολιτική για, την ε, βιομηχανική, για τη βιομηχανία που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχουμε και κάποιες κλαδικές πολιτικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να παρέμβουμε ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε επικίνδυνες τάσεις τις οποίες δεν έχει το περιθώριο να ε, κάνει η Ευρώπη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για την ε, ε σιδηροβιομηχανία και θα ήθελα να ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ε, υπάρχει το πρόγραμμα CARS 2020, αλλά θα θέλαμε και για τον τομέα της χαλιβουργίας ένα άμεσο πρόγραμμα δράσης. Θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε και τη δυνατότητα να έχουμε πολιτικές οι οποίες μας επιτρέπουν ε, να βοηθήσουμε τις στρατηγικές μας επιχειρήσεις ώστε να χαίρουν των καλύτερων δυνατών συνθήκων για να είναι ανταγωνιστικέ παγκοσμίω και να ε, είναι και καινοτόμε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνοδεύεται και με πολιτικές οι οποίες ε, μπορούμε, ε, τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε, έρευνα και καινοτομία δηλαδή, που αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και επίση θα ήθελα να σταθώ και στην ανάγκη να επανεξετάσουμε την πολιτική ανταγωνισμού, η οποία έχει σταματήσει από τη δεκαετία του 90 και δεν λαμβάνει πλέον υπόψη της τις απαιτήσει της ευρωπαϊκής οικονομίας, που είναι αντιμέτωπη με μια αγορά ε, παγκόσμιο ανταγωνισμού. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα στην ενιαία αγορά για να δούμε και τι γίνεται με το κόστος της ενέργειας και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε και τη δέουσα προσοχή στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει ίσως να αναρωτηθούμε και κατά πόσον θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο συμβούλιο το οποίο θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη χαλιβουργία ε, και να προσπαθήσουμε να κτίσουμε την ορμή που χάσαμε από το 2002. Ευχαριστώ. Ε, παρόλα, ε... Και τώρα ο λόγος στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ταγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Ο τομέας της χαλιβουργίας είναι ένας τομέας κλειδί για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Προσφέρει θέσεις εργασίας σε 360.000 ανθρώπους και φυσικά ο κύκλος εργασίας ανέρχεται στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατέχει θέση κλειδί στην κατασκευαστική αλυσίδα. Μετά από τις προσπάθειες που έγιναν για την αναδιάρθρωση ε, από τις απώλειες που είχαμε από τη δεκαετία του 80-90, η χαλιβουργία είναι μια δυναμική και ανταγωνιστική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, πάσχει από μια σειρά από προβλήματα. Σήμερα το 12% του χάλιβα που ε, πωλείται παγκοσμίω προέρχεται από τις ευρωπαϊκές χαλιβουργίε. Ε, οι δικέ μας βιομηχανίε καλύπτουν το 80% τη Ευρωπαϊκή παραγωγής και εξάγουν το μεγάλο ποσοστό ε, του παγκόσμιου προϊόντος δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει στασιμότητα στην περιοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σε συνδυασμό και με τις υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών αποτελεί πρόβλημα για όλες μας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Χάλιβα. Ένα πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, κυρίως ασιατικές χώρες, οι οποίες έχουν χαλιβουργία που παράγει με πολύ χαμηλότερο κόστος. Εξάλλου, Ακόμα και η ζήτηση προϊόντων χάλιβα από εξοκοινωτικές χώρες ε, είναι σε μείωση, όπως είναι και σε μείωση και ε, η ζήτηση για εισαγωγές. Οι τιμές ε, για την ενέργεια είναι από τις υψηλότερες παγκοσμίως και δυστυχώς, αν κάνουμε και μια αντιπαράθεση με τις τιμές της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι διπλάσια από ό,τι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από προβλήματα μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεσμεύτηκα και τήρησα αυτή τη δέσμευση δέσμευση την οποία ανέλαβα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ε, όταν συναντήθηκα με τα συνδικότητα ε, τα οποία συνέδευε και η πρόεδρος Περβάν Περές ε, σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου προκειμένου να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από το καλοκαίρι του 2013. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου και στο τέλος αυτής της πρώτης συνεδρίασης οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ο κλάδος, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων καθόρισαν τις βασικές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο τομέας της χαλιβουργίας. Ένα από τα σαφή μηνύματα που προκύπτουν είναι να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των στόχων των διαφόρων πολιτικών ώστε να προστατεύσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα στην Ευρώπη και τις προοπτικές εργασίες ε, με σκοπό να μην υπάρχει και ε, καθίζηση της αλυσίδας παραγωγής που θεμελιώνεται, που βασίζεται στη χαλιβουργία. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου και εκεί θα κάνουμε μια απόπειρα να εμβαθύνουμε στα θέματα τα οποία συζητήσαμε στην πρώτη συνεδρίαση και επαναλαμβάνω σκοπεύω να παρουσιάσω στο Σώμα των Επιτρόπων ένα πρόγραμμα δράσης πριν από τις θερινές διακοπές του 2013. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο Χάλιβας μπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί, διότι κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας, πρόκειται για μια κρίση η οποία δεν είναι διαρθρωτικής φύσεως, πρόκειται για μια κρίση η οποία έχει άμεση σχέση με την ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και επομένω ο Χάλιβας μπορεί τα επόμενα χρόνια να ε, ξαναποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιομηχανική μας πολιτική δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονό ότι στο κείμενο για την επαναβιομηχάνηση τη Ευρώπη εξετάζουμε κάποιου τομεί του οποίου θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και ίσω και με κάποιε προσπάθειε ε, από πλευρά καινοτομία και με χρηματοδοτική συνεισφορά ουσιαστική και από τον ιδιωτικό και τον ιδόσιο τομέα, τομεί ε, υψηλή ποιότητα, παραδείγματο χάρη τη ε, οι οικολογικές κατασκευές ε, και τα καθαρά αυτοκίνητα και ο τομέας ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, είναι ένας από τους βασικούς πελάτες της χαλιβουργίας. Ο χάλιβας λοιπόν εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία στόχο έχει όπως γνωρίζετε πολύ καλά και όπως παρουσίασα και σήμερα το πρωί στις ομάδες του Κοινοβουλίου αλλά και στο Συμβούλιο θα θέλαμε μέχρι το 2020 το 20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προέρχεται από, τον, ε, ε, από τη βιομηχανία. Πρέπει βεβαίως να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε και τεχνολογίες ε, πιο προηγμένες, ώστε από εκεί και πέρα οι παραγωγοί να μπορέσουν να αυξήσουν και τις δυνατότητες καινοτομία που διαθέτουν. Και το ίδιο είναι σημαντικό και για τον τομέα του Χάλιβα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε θούμε και εδώ στην καινοτομία. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν παρά τις δυσχέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καθόλου αποφασισμένη να εργαστεί ε, για τον τομέα αυτό. Ζήτησα και στον Επίτροπο Άντορ να συμμετάσχει σε όλες τις πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να επιτύχουν ε, τον αντικειμενικό μας σκοπό διότι δύο πράγματα θέλω να έχω στο επίκεντρο της δράσης μας. Καταρχάς, ε, να καθησυχάσουμε αυτή την κρίση η οποία θα μπορούσε ίσως και να επιδεινωθεί και να προβλέψουμε τις συνέπειες της κρίσης και με τον κλάδο και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και βεβαίως και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι όπως γνωρίζουν πολύ καλά η κυρία Σαρτόρη και η κυρία Μπερές ανέκαθεν καλούσα στις συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου και τις δύο κυρίες ως εκπροσώπους των δύο αρμοδίων επιτροπών ε, που ενδιαφέρονται για τη στρατηγική για τη χολιβουργία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρόληψη θεωρώ επίσης ότι είναι τα δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο εργασίας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ώστε να διασφαλίσουμε ένα μέλλον στον τομέα της χαλιβουργίας το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα λαμπρό μέλλον. Ε, πρέπει να εργαστούμε, χρειάζομαι τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν συνεργαστούμε με ευφυή τρόπο θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο στον οποίο πιστεύουμε όλοι μας και ο οποίος βρίσκεται και στην ουσία της ερώτησης που παρουσίασε η Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου. Απάντησα και θεωρώ ότι συμφωνώ απόλυτα με τους ε, στόχους και τις σκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλτών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, εξ ονόματος του ΕΛΚ, το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Φρανκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε ορισμένους τομείς η Ευρώπη πλέον δεν είναι ανταγωνιστική. Αυτό είναι γεγονός και οφείλουμε να το αποδεχτούμε, όχι όμως να το υφιστάμεθα. Θα πρέπει δραστικά να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το εξωτερικό για κλάδους τόσο στρατηγικούς όπως είναι η χαλιβουργία. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη τεχνογνωσία 200 ετών και πλέον ε, στις ε, τυχαίες εξέλιξεις αγοράς. Χρειάζεται επιγόντως ευρωπαϊκή επέμβαση. Και σας ζητώ επίσημα να μας πείτε ποια στρατηγική στρατηγική θα υιοθετήσετε για να εμποδίσετε ορισμένες κυβερνήσεις, βλέπετε η Γαλλική, ε, να ε, κάνουν αυτές τις ε, άγονε και αντιπαραγωγικέ δράσεις για να αποφύγουν τις μετακαταστάσεις. Ευχαριστώ. Ομιλητή, επόμενος ομιλητής εξ ονόματος ομάδος S&D είναι ο συνάδελφος κύριος Μπέρντ Λάγκε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, Βεβαίως και σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειες που καταβάλλεται να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία. Και θεωρώ σωστό ε, τις τάσεις που βλέπουμε και στη Χαλιβουργία ε, να μειώνονται απλώς οι θέσεις απασχόλησης και να κλείνουν τα εργοστάσια, δεν θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Διάβασα κάτι που δήλωσε ο πρόεδρος ε, του κλαδού ότι από τις 500 ε, χιλιάδες θέσεις εργασίας θα πρέπει να περικοπούν οι 100.000, 25% δηλαδή βαθιά το μαχαίρι. Ε, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε έτσι να το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτή η βασική βιομηχανία στην Ευρώπη θα σταθεροποιηθεί και θα δημιουργηθούν ε, προοπτικές ανάπτυξης. Είναι ε, βασικό θεμέλιο. Θυμηθείτε την ΕΚΑΧ ε, της Ένωσης που ήταν πάρα πολύ επιτυχής και στην πολιτική, την ερευνητική και στη διαρθρωτική για τη χαλιβουργία. Ένα τέτοιο μοντέλο θα πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει. Ε, ε, ε, ισομερείς κατά το 1 τρίτο εργαζόμενοι εργοδότες Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εργαστούμε στο μέλλον υπέρ της χαλιβουρίας και βεβαίως χρειάζεται και καινοτομία ακριβώς για να έχουμε πάρα πολύ ε, τους και ε, όλκιμους χάλιβες ε, που να ε, μας βοηθάει αυτό στην βιομηχανία μας και να είμαστε και ανταγωνιστικοί και σε λογικό κόστος. Έχετε λοιπόν την υποστήριξή μας σε αυτή την κατεύθυνση. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Ισαμπέλ Ντουράν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, να μην ξεχνάμε τους ε, εργαζόμενους Φλωράνς και τις Λιέζ. Οι πρώτοι περιμένουν τις προσδοκίες του εργοδότη και οι άλλοι αντιμετωπίζουν έναν επαρκές κοινωνικό σχέδιο. Σίγουρα ε, είναι ανεπαρκής η προσπάθεια. Σίγουρα πρέπει να επαναβιομηχανοποιήσουμε την Ευρώπη και εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι 6 Δεκεμβρίου, γιατί να μην έχουμε και μια πρωτοβουλία για τη χαλιβουργία πέραν του ερευνητικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Για συνεργασία των κρατών μελών, αντί να αφήνουμε στι μεγάλε επιχειρήσει χαλιβουργία ε, να κάνουν τον νόμο για τι θηγατρικέ του και να αποφασίζουν αν θα επιβιώσουν ή αν ε, θα κλείνουν. Ε, δεν θα πρέπει να παίζουν με τα πλεονεκτήματα που λαμβάνουν και να εκμεταλλεύονται και, τις, και τα φορολογικά μέτρα. Θα πρέπει να, γίνει, να μπει μια οργάνωση και θα πρέπει ε, οι ποσοστώσει ε, εμπορία εκπομπών ε, να, να, να χρησιμοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα μεγάλος πρωταθλητής αυτού του αποθεματικού είναι η Arcelor Metal αυτή που... Ε, ε, εξάρτησε την, ε, το άνοιγμα μια ε, υψηκαμίνου από την παροχή δικαιωμάτων εμπορία εκπομπών. Θέλουμε μια φιλόδοξη Ευρώπη, μια φιλόδοξη πολιτική και σίγουρα δεν θέλω μια πολιτική και μια Ευρώπη χωρί χαλιβούρια και θέλουμε ο χάλιβας αυτός να είναι πραγματικά Ευρωπαϊκό. Ομάδα των Πρασίνων, EFD, καλώ βήμα τον συνάδελφο κύριο Κούρσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η χαλιβουργία στην Ευρώπη διανύει μια κρίση, έλλειψη ανταγωνιστικότητα, αύξηση του κόστου παραγωγής εξαιτίας πληθώρα αποφάσεων από το ενεργειακό και το περιβαλλοντικό πακέτο ε, που μειώνει υπερβολικά τα καυσαέρια μέχρι το 2020. Μόνο στην Πολωνία έχουμε αύξηση των ανέργων κατά 200.000 ανθρώπους και επίσης αύξηση των τιμών της ενέργειας και μάλιστα σε μια χαλιβουργία στην Ευρώπη ε, θα απολυθούν 8.000 άνθρωποι και πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές, ε, πολλές χαλιβουργίες στην Πολωνία. Θα έχουμε μετεγκατάσταση στην Ουκρανία, στην Ινδία γιατί εκεί δεν ισχύουν ε, περιβαλλοντικές διατάξεις. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε γιατί ε, δυστυχώς ε, είναι αμφίβολα θα επιστρέψουν αυτές οι εταιρείες στην Ευρώπη. Και σίγουρα ε, η χαλιβουργία που είναι μεγάλος εργοδότης διανύει σημαντική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές μας ρυθμίσεις να μην οδηγήσουν αύξηση της μετεγκατάστασης και όλα αυτά προς όφελος της Σοβιετικής ε, Ένωσης και της Κίνας. Γκουε, το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Ζακί Ενάν. Για ένα μισή λεπτό. αυτή την ερώτηση βρισκόμαστε στην καρδιά της βασικής ευρωπαϊκής αντίφασης. Θα υπηρετούμε τους ανθρώπους, τις ανάγκες, θα χτίσουμε το μέλλον ή θα έχουμε προσκοληθεί ε, στα μερίσματα, στον ασίδωτο ε, ανταγωνισμό που βασίζεται μόνο στο ντάμπινγκ στην ανταγωνιστικότητα. Ε, η χαλιβουργία και ο χάλιβας είναι στα τα θεμέλια της Ευρώπης. Πάρα πολλοί κλάδοι αναπτύχθηκαν ε, αναζητώντας την πρόοδο και ε, οι άνθρωποι έχουν μια τεχνογνωσία απίστευτη στα αυτοκίνητα, στο σιδηρόδρομο, τα τρόφιμα, στις συσκευασίε, εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, πλούτος εκ των όνου για τα εδάφη μας και για τους λαούς μας. Ε, είναι θεμέλιο της Ευρώπης και διανύει μεγάλο κίνδυνο. Βαμπύρ έχουν πέσει οι χρηματαγορές ε, επάνω του για να καταστραφούν μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Θα χαθεί η τεχνογνωσία και θα καταστραφούν ζωές ε, χιλιάδων εργαζομένων. Η, υπόθεση της ε, πραγματικά είναι ε, στη Φλωράν, στη Λιέγη κλείνουν εργοστάσια. 37 δισεκατομμύρια ευρώ τα πήγαν στο Λουξεμβούργο για λόγους φορολογικούς. Ε, ε, κλείνουν εργοστάσια συνεχώς, κρατούν μόνο τα πιο αποδοτικά. Στην Ινδία διατηρούν τα εργοστάσια τα οποία βασίζουν στον υδρότα και στο αίμα των Ευρωπαίων τους οποίους μετά πετούν όταν δεν τους χρειάζονται μια γαλλική παροιμία λέει ότι ο χτίστης ε, στον τοίχο φαίνεται, στον τρόπο με τον οποίο χτίζει ένα τοίχο. Ε, εκεί ε, θα φανεί λοιπόν, από, εκ του αποτελέσματος θα κρυθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματο των μη εγγεγραμμένων το λόγο έχει ο συνάδελφο κύριος Ανδρέα Μέλτσα για μισό λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ύφεση και συγκυρία βαριά για τη χαλιβουργία, ακριβώ γιατί χαμηλώνει η ζήτηση από την αυτοκινητοβιομηχανία ε, στι χώρε τη Νότια Ευρώπη που στενάζουν από το χρέο. Επιπλέον, ε, είναι μεγάλε οι διακοιμάνσει και στο κόστο τη ενέργεια και στι πρώτε ύλε και αυτό είναι πολύ δύσκολο για τη χαλιβουργία. Γι' αυτό ε, ε, συμπαρασύρεται και ο κλάδος ε, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης στα παλιοσίδερα. Ε, έχουμε ανταγωνιστές παγκοσμίω εκτός της Ευρώπης που δεν έχουν υψηλό κόστος ενέργειας, περιβάλλοντος και ε, πιστοποιητικών διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό έρχεται ο φθηνός χάλιβας όλο και περισσότερο και διεισδύει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς γιατί δεν έχουν αυτές τις βαριές προϋποθέσεις οι άλλοι. Θα πρέπει να το έχει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ε, που ε, μειώνει τις άδειε και τα πιστοποιητικά και αυξάνει το κόστος του διοξίδιου του άνθρακα. Ακούμε λέει ότι θα καταργηθούν το 1 τέταρτο των θέσεων εργασίας και των δυνατοτήτων. Πώς θα γίνει αυτό. Μακροπρόθεσμα σημαίνει ότι μέχρι το 1 τέταρτο των εργαζομένων, δηλαδή 100.000 θέσει εργασία θα καταργηθούν. Αν συμβεί πραγματικά αυτό, ε, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει ενεργά και γενναία για να αντιμετωπίσει την οικονομική και κοινωνική συνέπεια. Οι άλλοι εγγεγραμμένοι το λόγο έχει Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο κυρία Σαρτόρη διότι ζήτησε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ο τομέας του Χάλιβα, ο οποίος είναι θεμελιώδης για το ευρωπαϊκό σύστημα, ε, ζει μια καθίζηση με απώλεια θέσεων εργασίας. Πρώτο πρόβλημα, οι ε, εισαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κίνα είναι ο πρώτος ε, προμηθευτής, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι χώρες αυτές παράγουν σε συνθήκες του ανταγωνισμού, έχουν ακατάλληλους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κανόνες είναι λιγότερο δεσμευτικοί ε, για τι κρατικέ ενισχύσεις και είναι πολύ πιο χαμηλό το κόστος της ενέργειας. Κύριε Επίτροπε Ταγιάννη, βεβαίω ε, ε, εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τη στρατηγική για τον τομέα του Χάλιβα, τον οποίο ετοιμάζετε και σας ευχαριστώ διότι επανειλημμένω είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικαιροποιήσει του κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει και τον ανταγωνισμό. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θα ήθελα να σταθώ ε, στο Τέρνη. Η περιοχή του Τέρνη είναι βιομηχανική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο ιταλική ε, κληρονομιά. Είναι από τους πρώτους παραγωγούς ε, για τα ανοξίδωτα. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλος έλεγχος της ποιότητας, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα σε θέματα ρήπανσης και ανακύκλωσης και ε, το κοινοτικό αντιτρός ε, το οποίο είναι κατά του μονοπωλίου ε, διακήρυξε ότι η περιοχή του Τέρμη είναι ε, ε, ε, ακατάλληλο και άφησε τη δυνατότητα παραγωγής στη Φιλανδία. Παρήγαγε πάρα πολλές θέσεις εργασίες και χωρίς αυτή τη δυνατότητα ε, χάνει την ανταγωνιστικότητά της η περιοχή και δεν θα υπάρχει και ενδιαφέρον από τους πιθανούς αργωνιστές. Γι' αυτό ακριβώς είναι ανησυχητικά τα ζητήματα. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε λοιπόν ότι θα έχουμε βιομηχανικά προγράμματα μακροπρόθεσμα, ανταγωνιστικά που θα καθορίζει ότι θα έχουμε κατάλληλους κανόνες αγοράς και θέματα απασχόλησης στρατηγικές πρέπει να λάβουμε για το κόστος τη ενέργεια. Γιατί να μην υπάρχει μια πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων ε, χάλιβα. Ευχαριστώ πολύ. Λίλη, Ιταλικής παρουσίας συνέχεια. Το λόγο έχει η συνάδελφο κυρία Πατρίτσια Τόγια για 1,5 λεπτό. Grazie. Ευχαριστώ. Η ενεργειακή κρίση ε, κάνει ε, να πληρώσουμε ένα πολύ ακριβό το τίμημα για τις θέσεις απασχόλησης, έχουμε επισφαλείς θέσεις εργασίας ε, και προσωρινές εργασίες του συγκεκριμένου τομέα. Πολλές φορές ε, όλοι στρέφονται προς την από Ανατολή και στις Ηνωμένε Πολιτείες για την παραγωγή. Και εδώ ανησυχούμε για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν εμείς ως Ευρώπη να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε καλύτερη βασική παραγωγή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να προστατεύσουμε το συγκεκριμένο τομέα. Θα σας υποστηρίξουμε κύριε Επίτροπη αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο που έχουμε λάβει σε θέματα βιομηχανίας. Και επίσης θα ήθελα να πω και κάτι για τις ε, διτές θέσεις που ακούγονται. Όχι σήμερα, αλλά πολλές φορές υπάρχει μια ε, διπλή στάση ε, ξεχωριστή για το περιβάλλον και ξεχωριστή για τις θέσεις εργασίας. Ένας βιομηχανικός κλάδος λοιπόν που θεωρείται χαλιβουργία αναπόσπαστο τμήμα του θα πρέπει να έχει προηγμένες τεχνικές, λύσεις που θα καθορίζουν τα διάφορα συμφέροντα και τις διάφορες απαιτήσει. Γι' αυτό και ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε σημαντικό σχεδιασμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα πρέπει πρέπει να οπισθοδρομήσουμε κατά την άποψή μου, διότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε νέε τεχνολογίε, νέε διαδικασίε, ε, πιστοποίηση των εγκαταστάσεων για να έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά του πόρου του και του ενεργειακού τη πόρου και μάλιστα με φαλτήριο του ενεργειακού πόρου θα πρέπει να αναζητούμε και νέε πηγέ ε, βιομηχανία. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος κυρία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Πολωνία έχουμε περιοχές όπου οι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους και ενώ οι εργοδότες τους ε, εισάγουν ε, φθηνό χάλιβα από την Κίνα. Αυτό είναι χαρακτηριστική περίπτωση διαφυγή διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή το πρόβλημα της εμπορίας των εκπομπών θα αναλάβει κάποια μέτρα γιατί είναι ανησυχητική η κατάσταση. Και το backloading που προτείνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη χαλιβουργία σήμερα. Γιατί επηρεάζει μια τέτοια απόφαση όχι μόνο τις τιμές αλλά ξέρουμε ότι το backloading είναι το πρώτο βήμα για διορθωτικές παρεμβάσεις σε τα site και αντίστοιχα μέτρα. Ε, επίσης, θέλουμε κάποιες καθυστερήσεις με γραμμές για κάποιες κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να αντισταθμιστούν ε, τα, τα κόστη. Γιατί δυστυχώς ε, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, χρήματα για να δώσουν αυτές τις αποζημιώσεις. Επίσης έχουμε και το σχέδιο για την COP, τη 18η ΚΟΠ. Έχουμε όλο και αυξανόμενο ποσοστό εισαγόμενων εκπομπών. Θα πρέπει στα πλαίσια των δράσεών μας να είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις μας θα είναι αποτελεσματικές και να μην εξαγάγουμε θέσεις εργασίας προκειμένου να εισαγάγουμε μόλυνση του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ο μιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Ρομπέρτο Γουαλτιέρη για λεπτό. Μάικρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι παρούσες δυσκολίες της χαλιβουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιτάσσουν να λάβουμε υπόψη μας το ρόλο της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες ε, στην ε, βιομηχανική πολιτική, αλλά θα πρέπει να δούμε και συνολικά τι γίνεται με τις πολιτικές ανταγωνισμού, τις φορολογικές και ούτω καθεξής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε τις στάσεις μας, διότι στο παρελθόν είχαμε μία τοποθέτηση που στο παρελθόν ευνοούσε την κατανάλωση ε, και ε, άλλα ωφέλη και όχι τη βιομηχανία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ε, βιομηχανίες όπως ε, η χαλιβουργία στο Τέρνη και ε, στο Πιομπίνο και δείχνουν ότι πρέπει να λάβουμε επιτακτικά μέτρα. Θα πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια αξιολόγηση και όχι μόνο ευρωπαϊκή για να δούμε ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις και από εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ακέραιη η περιοχή του ε, σε αυτή τη διαδικασία παροπλισμού που γίνεται, που ε, γίνεται και να δούμε και τι γίνεται και με την Υψικάμινο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ε, και τα όσα περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Ανάπτυξης του Ιουνίου που είναι υπέρ πολιτικών ε, δημοσιονομικής εξηγίανσης υπέρ της ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα αυτά. Επίσης, το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Μπορεί να χρειάζεται να δώσουμε και βοήθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια στην παραγωγή για μεγάλη στρατηγική σημασία χαλιβουργία. Ευχαριστώ. Ε, στο βήμα την κυρία για δύο ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά σπαράζει η καρδιά μου όταν βλέπω να κλείνουν σιγά σιγά και σχεδόν μοιραία όλες οι μονάδες ε, ε, παραγωγής της χαλιβουργίας του Σεφλάνς που είναι η γερέτη ράμου. 70 είναι ακόμα οι εργαζόμενοι, ενώ στην αρχή της δεκαετίας του 80 είχαμε 3.000 ε, μισοτού που έκαναν αυτή τη ε, ε, μονάδα να ζει, φεύγει, χάνεται ένα τμήμα ιστορίας όσο και μνήμης και πραγματικά θλίβομαι πάρα πολύ μαζί με τους συμπολίτε, όσο και εξοργίζομαι και εδώ και αλλού. Ωστόσο δεν συμφωνώ ότι οι κακοί καπιταλιστές κλείνουν τα εργοστάσια για να ε, θρέψουν αρκετά ε, παχύσαρκους ήδη ε, μετόχους. Είναι μεγάλη η παραγωγή αλλά και πολύ μεγάλη η ευρωπαϊκή φρενίτιδα η κανονιστική και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτά είναι πραγματικά ε, αναμφισβήτητα. Και εγώ δεν κατηγορώ εκείνους που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Απλώς ε, ε, οι συνέπειες του κλεισίματος των εργοστασίων είναι ολέθριες. Χάνονται όχι μόνο θέσεις εργασίας αλλά και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και θα πρέπει να αντιδράσουμε όχι με φρούδες υποσχέσεις αλλά μπαίνοντα δεσμευτικά στο δρόμο μιας βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη που να αξίζει το όνομά της. Έχουμε στρατηγικά συμφέροντα να υπερασπιστούμε πιστούμε στην Ευρώπη. Και η χαλιβουργία είναι οπωσδήποτε ένα στοιχείο βιομηχανικής πολιτικής πάρα πολύ σημαντικό. Ε, βιομηχανική πολιτική, προσέξτε, δεν σημαίνει προστατευτισμός ή κλείσιμο συνόρων. Αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι ε, και ε, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Μας το δείχνουν οι εταίροι μα το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και στη Χαλιβουργία θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα ορισμό ελάχιστων κανόνων για να μην ε, σκοτώσουμε μια βιομηχανία που θα, φύγει, που θα ξαναρχίσει μάλλον ε, να αναπτύσσεται όταν περάσει αυτή η συγκυρία. Αυτά που συμβαίνουν όμως είναι οριστικά και η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική ε, θα μπορούσε να ε, απαντήσει χωρίς να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στους εταίρους και ανταγωνιστές μας. Νομίζω κύριε Επίτροπε ότι καταλάβατε το μήνυμα, αλλά χρόνο πια για χάσιμο δεν έχουμε. Η κυρία Λούλινγκ με συνδέει σχέση καλής γειτονίας στη χωροταξία της Ολομελίας. Εξού και η επίοικια την οποία επέδειξα ως προς το χρόνο. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Φρεντερίκ Νταρντέν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η χαλιβουργία είναι ένα τομέα του μέλλοντο. Είναι περί τώρα παραλάβουμε. Οι εργαζόμενοι στον κράτο αυτό έχουν αναπτύξει μια πραγματική τεχνογνωσία. Και η πρώτη ύλη τη χαλιβουργία είναι σημαντική και για την αυτοκινητοβιομηχανία. Και εκεί έχουμε σημαντικό τμήμα του οικονομικού μα ιστού. Γι' αυτό και έγιναν και πολύ σημαντικέ επενδύσει, πολύ συχνά με την ε, συμμετοχή και δημοσίων κονδύλιων για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη νέων χαλιβουργικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αλλά α πάρουμε ένα παράδειγμα που χαρακτηρίζει τι παρεκτροπέ των μεγάλων ομάδων. Εδώ και πολλά χρόνια η ArcelorMittal ε, στη Μοζέλη, το Λουξεμβούργο, τη Λιέγη, εφαρμόζει μια στρατηγική σταδιακή καταστροφή του κεφαλαίου παραγωγή τη. Ποια είναι τα θεμέλια τη στρατηγική τη. Ο Όμιλο κλείνει ε, βιώσιμα και αποδοτικά εργοστάσια, χρησιμοποιώντα τον ανταγωνισμό μεταξύ του για να επαναπροσανατολίσει τι επενδύσει του και απορρίπτει την ιδέα να παραχωρήσει ε, τις, τα βιώσιμα εργοστάσια προκειμένου σε έναν ανταγωνιστικό κο εταίρο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπίσουμε τους κανόνες ε, του υγιούς και θεμητού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ε, δεν είναι καταχρηστική πολιτική το να εμποδίσουμε μια εξαγορά. Δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί και με την περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ένα λεπτό. Merci, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Είχαμε τρει αλλεπάλληλε συζητήσει σήμερα σχεδόν στην ημερήσια διάταξη. Βρίσκεστε στην καρδιά τη συζήτηση και μάλιστα μερικές, σε μερικέ συζητήσει πρωτοστατήσατε από κοινού με τον Επίτροπο Άντορ. Ε, γιατί μιλούμε για τη βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική που βρίσκεται στην καρδιά και των Ευρωπαίων. Αλλά λείπει ένα σημαντικό παράγοντα από τη συζήτηση, ο Επίτροπο Μπαρνιέ. Γιατί βλέπουμε ότι πίσω από πολλέ στρατηγικέ ε, κρύβεται η χρηματοδότηση μια οικονομία ε, που όμω ξυλώνει το βιομηχανικό ιστό στι περιοχέ μα. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο να ξαναρχίσουμε να χτίζουμε αυτό το νηστό. Χαιρόμαστε για πρωτοβουλίες που ακολουθούν μια, ένα λογικό ήρμο μεταξύ της επιχειρηματολογίας για τις πρώτες ύλε και της επιχειρηματολογίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλουμε μια σφαιρική στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης με εμβρόντιτη απέναντι στην κινητοποίηση των Ευρωπαίων και στην έλλειψη πρόσβασης ε, στις σπάνιες γέες, ε, ενώ είναι στρατηγικό το θέμα και ε, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό οι Αμερικανοί. Και όταν μιλούμε για τη χαλιβουργία στους Ευρωπαίους, δεν τη σαν να μην τη θεωρούν στρατηγική σημασία για τις οικονομίες. Και αφήνουμε τον κύριο Μιτάλ να συμπεριφέρεται ως ε, ε, οικονομολόγος και ε, ουσιαστικά καταπατάει όσα μάθαμε στα βιβλία της οικονομίας. Αντί να δημιουργεί προσθεθέμενη αξία, καταστρέφει μονάδες παραγωγής σε, στην Ευρωπαϊκή Έδωση για να οργανώσει καλύτερα την κερδοσκοπία. Ευχαριστώ. Ε, ανοίγει η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑ. Υπάρχουν τρεις αιτήσει ε, Θέλετε και εσείς κύριε Παλώνε. Ο κύριος Παλώνε έχει... No, Ο κύριος Παλώνε έχει... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά λακωνικός. Δύο ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Ταγιάννη. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό, με κάποια άλλα διαφωνώ. Όσον αφορά όμως τη στρατηγική σημασία της χαλιβουργίας ε, στην Ευρώπη, συμφωνώ. Συχνά όμως ε, καθόμαστε και με ψημιρούμε και δεν ε, βλέπουμε, κύριε Ταγιάννη, ότι ο κόσμος άλλαξε. Όταν μιλάμε, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, για κυρίαρχη θέση, κυρίαρχη θέση σημαίνει να δούμε τι γίνεται με τα θέματα αυτά δεσπόζουσα θέση. Το 1880 ο κόσμος ήταν διαιρεμένος στα δύο. Απ' τη μία είχαμε την Ευρώπη και απ' την άλλη είχαμε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα ο κόσμος άλλαξε. Έχουμε τελείως διαφορετικές ε, καταστάσεις, έχουμε νέες αγορές, την Ινδία, την Κίνα, τη Βραζιλία και επομένως ε, υπάρχει μεν ε, ανταγωνισμό σε κάποιες περιπτώσεις αθέματος, αλλά πρέπει να αλλάξουμε την παλιά νομοθεσία που είναι παροχημένη πλέον. Και επίσης πότε θα γίνει αυτή η ευλογημένη συγχώνευση, τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Σαρτόρη, διότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας μας επιτρέπει επιτέλους να συζητήσουμε ε, τα συμφέροντα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Χάρη στα συμφέροντα τα οποία οθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στην ε, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και να λαμβάνει μονόπλευρες πολιτικές, κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους οι χαλιβουργίες επειδή ακριβώς είναι ενεργοβόρες βρίσκονται σε πιο δινή θέση σε σχέση με τις ε, υπόλοιπες ε, βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ε, τις ποσοστώσεις που τους δίνονται για την ενέργεια και χάνουν και τις δυνατότητες να μπορούν από εκεί και πέρα να αγοράσουν δυνατότητες σε αυτό το θέμα. Το 2011 έχασαν το 10% της αγοράς και το, για το 2012 προβλέπεται ότι θα χάσουν ένα 12% ακόμα μεριδίου της αγοράς. Η μόνη λύση λοιπόν για να αποφύγουμε τον αθόμητο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες είναι να επιβάλλουμε δασμός ε, στα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία θα είναι ανάλογα με την παραγωγή ε, σε σχέση με τρίτες χώρες. Στη διαδικασία ο συνάδελφος κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Ταγιάννη, χθε το απόγευμα μια ολόκληρη πόλη στην περιοχή μου, στην Τοσκάνη, σταμάτησε για δύο ώρε. Δέκα χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στου δρόμους, εργαζόμενοι, έμποροι, ε, άνεργοι, απλοί πολίτε. Ε, έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και εγώ θα ήθελα να κάνω το ίδιο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πόλη κινδυνεύει να πεθάνει διότι κινδυνεύει ο τομέας της χαλιβουργίας όπου το πιο μπίνο ζει εδώ και δεκαετίες. Ε, κινδυνεύουμε να έχουμε χιλιάδε θέσει εργασία χαμένε και φυσικά θα υπάρχουν συνέπειε και στην καθημερινότητα των πολιτών αυτών. Θέλουμε λοιπόν να αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα για να διασώσουμε την Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία η οποία αντιμετωπίζει τεράστιε δυσκολίε και τιμωρείται από τεράστιο ανταγωνισμό κυρίω από την Κίνα. Από το Χάλιβα το 1951 ξεκίνησε η οικοδόμηση της Ευρώπης, την Ευρώπη την οποία, στην οποία ζούμε σήμερα και επομένως είναι κρίμα ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην δρούν για να προασπίσουν το συγκεκριμένο τομέα, ο οποίο θα πρέπει να θεωρείται ακόμα στρατηγική σημασία και προτεραιότητα. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαφώς οι παρεμβάσεις όλων των Ευρωβουλευτών που έλαβαν το λόγο σήμερα στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού συστήματος. Ο τομέας του Χάλιβα, όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, απαντώντας ε, στην ερώτηση της κυρίας Σαρτόρη, αποτελεί στοιχείο κλειδί. Ο ανταγωνισμός βέβαια τη σήμερα ημέρα στον κόσμο σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε και μια πραγματικότητα η οποία είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, όπως άλλωστε είπαν αρκετοί από τους ευρωβουλευτές ε, στη διάρκεια της σημερινή συζήτηση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τόσο και στη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας ε, συζητήσαμε το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής ε, και την ισχύ που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο και τι προβλήματα αντιμετωπίζονται σε ένα πλαίσιο το οποίο επαναλαμβάνω ότι έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που είχαμε στη δεκαετία του 50 και η συζήτηση συνεχίζεται και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έλαβα και μια σχετική επιστολή από 7 χώρες οι οποίες ε, είναι οι βιομηχανοποιημένες χώρες, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση επί του ζητήματος και στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Ο Επίτροπος Αλμούνια, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την πολιτική ανταγωνισμού σκοπεύει να παρουσιάσει ένα σχέδιο μεταρρύθμισης. Η συζήτηση συνεχίζεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι πρέπει να συμβαδίζουμε με τους καιρούς μας. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κανόνες ε, του ανταγωνισμού είναι θεμελιώδης σημασία για την ανάπτυξη και δεν μπορούμε να προασπίσουμε την ενιαία αγορά ε, χωρίς αυτούς. Νομίζω ότι αυτό ακούσαμε από όλους τους ευρωβουλευτές και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και θα πρέπει να το εξετάσουμε τους επόμενους μήνες εάν θέλουμε να έχουμε ένα βιομηχανικό σύστημα ανταγωνιστικό. Και για να απαντήσω και στην κυρία Περβάνς ε, Περές και η πολιτική της ενίας αγοράς ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την περίπτωση. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ είναι υποστηρικτής, ένθερμος υποστηρικτής μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής και πάντα με στήριζε για όλες τις πρωτοβουλίες ε, τις οποίες ε, θέλησα να προωθήσω, συμπεριλαμβανομένες και της πολιτικής για τη χαλιβουργία. Θεωρώ λοιπόν ότι σε πολιτικό επίπεδο σαφώς υπάρχει βούληση. Επιμένω για το, αυτό το στόχο του 20% διότι ε, πέραν του 20% για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει και το 20% του ΑΕΠ το οποίο θα σχετίζεται με τις βιομηχανικές πολιτικές σαφώς ε, εκκρεμούν πολλά πράγματα στον τομέα του Χάλιβα. Ε, υπάρχει το θέμα του, ε, της χαλιβουργίας στο Τέρμι, το οποίο έθιξαν αρκετοί συνάδελφοι και να πω ότι έγινε, έδωθηκε μια απάντηση ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις αποζημιώσεις. καταφέραμε να έχουμε ε, υψηλό ποσοστό για τις κρατικές ενισχύσεις στο, στο συγκεκριμένο τομέα και σε όλους τους τομείς ε, έχουμε συμπεριλάβει ε, και τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους όπως επίσης και την χαλιβουργία. Όσον αφορά τώρα το backloading, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία πρόταση ε, με τη στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μπορεί να μας δώσει και την άποψή του, διότι χωρίς τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο συγκεκριμένο τομέα. Σημειώνω βεβαίως τις ανησυχίες ε, των ε, προβουλευτών, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε διότι νομίζω ότι γίνεται να συγκεράσουμε την εμπορική και την βιομηχανική πολιτική. Και για να απαντήσω και στην κυρία Ντουρά. Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για το ορίζοντα 2020 θα εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή έρευνα προκειμένου να έχουμε πιο αποτελεσματική παραγωγή και απόψη πόρων και απόψη ενέργειας και η χολιβουργία μαζί με άλλους κλάδους ε, ήδη έχουν υποβάλει πρόταση για μια νέα εταιρική σχέση και σύμπραξη ε, ε, τομέα που λέγεται SPIRE. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά και στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, το οποίο έφυξα και εγώ, αλλά στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Μέτσλερ στην παρέμβασή του και το υπενθύμασε και η κυρία Περβάν Περές, θα πρέπει να εξετάσουμε ε, το θέμα αυτό όχι ως το μόνο πρόβλημα που υπάρχει. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια στρατηγική για τις πρώτες ύλε και για τον τομέα του Χάλιβα. Όπως γνωρίζετε έχουμε υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες με εξοκοινωτικές χώρες και ε, ξεκίνησε και η εταιρική σχέση για την καινοτομία για την ε, ανακύκλωση και την εξόριξη πρώτων υλών. Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή πολιτική που θα χρηματοδοτηθεί και από τις παρούσες και τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεσμεύεται ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσον αφορά τώρα το τέρνη, θεωρώ ότι ο Επίτροπος Αλμούνια έδρασε σεβόμενος πλήρως ε, τους ισχύοντες κανόνες το γεγονός ότι έμεινε ενωμένο το βιομηχανικό ε, σκέλος του Τέρνη είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο μπορεί να μας επιτρέψει την πώληση του συγκεκριμένου εργοστασίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Θα ήταν επιζήμιο να είχε κατακαιρματιστεί. Το να είναι ενωμένο σημαίνει ότι μπορεί να απολυθεί στην αγορά με καλύτερες εγγύησεις τόσο όσον αφορά την προστασία της ίδιας της εγκατάστασης όσον αφορά και την προστασία ε, της, ε, των θέσεων εργασίας. Ε, όσον αφορά τώρα την Υψικάμινο, όντω αυτό δεν ε, ε, αφορούσε το σύνολο της, ε, του εργοστασίου. Οι ιδιοκτήτες όμως είναι διατεθειμένοι να απολύσουν και αυτό το τμήμα. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και το πρόβλημα το οποίο ανέφερε η κυρία Αλτζελίλη θα μπορούσε να επιληθεί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτή την σημαντική βιομηχανική περιοχή και για την Ιταλία, που είναι σημαντική και για την Ιταλία αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το ξανασυζητήσουμε άλλωστε στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 10 ε, Δεκεμβρίου. Ένα Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, στο οποίο θα δοθεί περισσότερη σημασία στην ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανικής πολιτικής και των εκπροσώπων της βιομηχανίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κυπριακή Προεδρία για τη βοήθειά της ε, στη συγκεκριμένη δράση. Ε, στις 9 του μηνός το βράδυ σκοπεύω να συναντήσω και τους ε, υπουργούς βιομηχανίας για να συζητήσουμε και το θέμα της κρίσης της αυτοκινητοβιομηχανίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κρίση της χαλιβουργίας. Από πλευράς λοιπόν Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το βιομηχανικό μας σύστημα, να γίνει ένα πιο σύγχρονο, πιο ανταγωνιστικό, πιο συμβατό σύστημα, αλλά σαφώς θα πρέπει να αποτελέσει και έναν από τους σημαντικούς μοχλούς για τη διέξοδο από την κρίση και την προστασία των θέσεων εργασίας είμαι απόλυτα πεπισμένος και ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε ότι οι θυσίες τις οποίες ζητήσαμε από τους συμπολίτες μας είναι απαραίτητες αλλά όταν οι θυσίες δεν συνοδεύονται και από μια ισχυρή πολιτική ανάπτυξη και συνεπώς και από μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική, ου μόνον ελοχεύει ο κίνδυνος να είναι άχρηστες, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος και να είναι και επιζήμιες για τους συμπολίτε μας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εργαστούμε και στα δύο μέτωπα και είναι και ευθύνη μου αλλά και βούλησή μου να υποστηρίξω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική ανάπτυξη φροντίζοντας ε, να γίνει και πιο ανταγωνιστικός ο τομέας της χαλιβουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση κυρίστε περιομένη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Κομισιόν με θέμα προσεχή παγκόσμια διάσκεψη για τι διεθνεί τηλεπικοινωνίε τη Διεθνού Ένωση Τηλεπικοινωνιών και ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών.